Rebonjour, Καλησπέρα σας και πάλι. Ευχαριστούμε που είσαστε εδώ για τη δεύτερη ενημέρωση την Επιτροπή σήμερα. Έχουμε τον Επίτροπο Αβραμόπουλο μαζί μας, ο οποίος θα σας ενημερώσει για ένα σημείο που ανέκρινε το Συμβούλιο νωρίτερα σήμερα, συστάσεις για τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα. Έχετε το λόγο, Επίτροπε. Thank Ευχαριστώ, Μαργαρίτη. Καλησπέρα σας. Ξέρω ότι ήσασταν πολύ απασχολημένοι σήμερα. Ξέρετε ότι τους τελευταίους μήνες έχουμε λάβει σημαντικά βήματα για να ενισχύσουμε και να βελτίσουμε τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα βοηθήσει να επανέλθει ο χώρος Σέγγεν στην ε, κανονική του λειτουργία. Να είμαι απόλυτα σαφή, η πρώτη μα προτεραιότητα ήταν και παραμένει η διαφύλαξη του Σέγγεν, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα τη Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Όλε μα οι προσπάθειε ε, στοχεύουν προ αυτόν τον τελικό στόχο. Να επανέλθουμε σε μια φυσιολογική λειτουργία τη περιοχή Σέγγεν χωρί εσωτερικού ελέγχου τάχιστα, όσο πιο γρήγορα γίνεται. Γι' αυτό ήταν τόσο κρίσιμη σημασία η έναξη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή και Συνοριοφυλακή. Τώρα λοιπόν πρέπει να λειτουργήσει φυσιολογικά. Αυτό έχει θεμελιώδη σημασία, αλλά δυστυχώ δεν έχουμε φτάσει ακόμη σε αυτό το σημείο. Πριν από μερικέ εβδομάδε, όταν κάναμε την διάμεση έκθεσή μα, ανέφερα ότι οι έλεγχοι μέχρι στιγμή ήταν αναγκαίοι και ε, σέβονται την αρχή τη αναλογικότητα. Η Κομισιόν παρακολουθεί την κατάσταση από πολύ κοντά θέλω να πω σαφώς ότι έχουμε πλήρη συνέστηση όλων των ανησυχιών και των κρατών Σέγγεν που ακόμη διεξάγουν εσωτερικούς ελέγχους να συμπεθυμίσουν η Γερμανία, Αυστρία, Σουηδία, Δανία και Νορβηγία και οι γείτονοι, οι γειτονικές χώρες του Σέγγεν που δεν το κάνουν μετά το αίτημά μας οι πέντε χώρες Σέγγεν αυτές μας έδωσαν στοιχεία όπου βλέπουμε ότι έχουν μειωθεί οι αφήξεις και οι αιτήσει ασύλου που έχουν υποβληθεί. Όμως οι εξαιρετικές ε, περιστάσεις που ιδεολόγησαν την εισαγωγή των εσωτερικών ε, συνοριακών ελέγχων εξακολουθούν να ισχύουν. Πρώτον, μια σειρά από παράτυπους ε, μετανάστες, πολλοί 60.000 περίπου, εξακολουθούν να είναι στην Ελλάδα και θα έπρεπε να μετακινηθούν προς άλλα κράτη-μέλη εάν, μετακιν... καταργηθούν αυτές οι εσωτερικοί έλεγχοι. Δεύτερον, υπάρχει αρκετή πίεση ε, επί των υπηρεσιών ασύλου των πέντε χωρών Σέγγεν μετά τον αριθμό αιτήσεων ασύλου που έλαβαν και αυτών που επίκυνται επιπλέον. Ορισμένα στοιχεία που είχαμε εντοπίσει στον οδικό χάρτη μας για την επιστροφή στο Σέγγεν θέλουν περισσότερο χρόνο για να εφαρμοστούν πλήρως και με βιώσιμο τρόπο. Ελπίζω ότι σε τρεις μήνες ότι θα λειτουργεί πλήρως η Ευρωπαϊκή Άκτο και Σύνοριο Φυλακή και συνεχί, ε, θεωρούμε ότι θα συνεχίσει να ισχύει με βιώσιμο τρόπο η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και εργαζόμαστε για να επιτύχουμε την πλήρη εφαρμογή των κανόνων του Βερολίνου ανεξάρτητα από οποιαδήποτε περαιτέρω μεταρρύθμιση. Ενώ συνεχίζουμε να ε, θέλουμε να υπάρξουν αποτελέσματα για την επίτευξη των στόχων μετεγκαταστάσεων. Γι' αυτό η Επιτροπή προτείνει να παραταθεί το καθεστώς των εσωτερικών συνοριακών ελέγχων στα ίδια σημεία ε, των συνόρων μας, αλλά τονίζω για μία αυστηρά περιορισμένη περίοδο ενός επιπλέον τριμήνου. Αυτή η περιορισμένη παράταση που προτείνουμε στοχεύει στην προσαρμογή των ε, υπαρχόντων προσωρινών ελέγχων, ούτως ώστε να ανταποκρίνονται στις υπάρχουσες ανάγκες. Δηλαδή οι έλεγχοι θα πρέπει να διεξάγονται μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίοι και πρέπει να είναι περιορισμένοι στην έντασή τους στο απόλυτα ελάχιστο απαιτούμενο. Αυτό σημαίνει ότι ε, εάν για κάποια περίοδο δεν υπάρχουν ε, αξιοσημείωτες ροές. Κάποιοι έλεγχοι για ορισμένα τμήματα των συνόρων μπορεί να μην είναι πλέον αναγκαίοι. Θέλω να είμαι σαφής ότι αυτό που προτείνουμε σήμερα είναι η εξαίρεση για εξαιρετικές περιπτώσεις. Δεν είναι το νέο φυσιολογικό. Γι' αυτό τονίζουμε και απαιτούμε η αναγκαιότητα αυτών των ελέγχων να επανεξετάζεται τακτικά σε συνεργασία με όλα τα κράτη-μέλη που εμπλέκονται και με στόχο σταδιακής μείωσής τους. Ζητάμε από τα κράτη-μέλη να υποβάλουν ε, μηνιαίες ε, εκθέσεις καθώς και μία αποτίμηση για την συνεχιζόμενη αναγκαιότητα αυτών των ελέγχων. Όλες μας οι προσπάθειες και η σημερινή πρόταση έχουν μόνο ένα στόχο να αντιμετωπίσουμε περαιτέρω όλες τις προκλήσεις για το μεταναστευτικό και την ασφάλεια για να καταργηθούν όλοι αυτοί οι εσωτερικοί έλεγχοι όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Έχουμε ε, οικονομικές εκτιμήσεις για το κόστος ε, της ε, κατάργησης του Σέγγεν, αλλά το κοινωνικό κόστος θα ήταν πολύ μεγαλύτερο, αν όχι δυσθεώρητο. Η Κομισιόν και εγώ προσωπικά Είμαστε απόλυτα και σταθερά δεσμευμένοι για να διαφυλάξουμε αυτό το σοβαρό ευρωπαϊκό κεκτημένο που δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο και ε, να μην παρερμηνευθεί η σημερινή μας πρόταση. Δεν θεωρούμε ότι είναι δεδομένο. Αντίθετα, είμαστε αποφασισμένοι να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη για να επανέλθει το Σέγγεν στην κατάσταση που θα έπρεπε να είναι. Ελεύθερη εσωτερική κυκλοφορία των ατόμων χωρίς ελέγχου στα σύνορα με ισχυρή διαχείριση των εξωτερικών μας σύνορων. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Έχουμε τώρα το υλικό για τον τύπο που έχει κυκλοφορήσει εδώ στην αίθουσα και έχει τυπωθεί και όλες. Υπάρχει χρόνος για ερωτήσει, Παρακαλώ. Νταβίτ Καρέτα από το από το Ιταλικό ραδιόφωνο. Εδώ είμαι, Επίτροπε. Δύο ερωτήσεις, αν επιτρέπετε. Η πρώτη, για τους 60.000 μετανάστες στην Ελλάδα. Είπατε ότι θα μπορούσαν να μετακινηθούν σε άλλα κρατημέλη. Όμως ε, αυτός ο κίνδυνος θα επικρέμεται για πάντα βάσει των κανόνων πόσο θα μείνουν στην Ελλάδα. Γιατί το, ζήτημα αρχίζει να παλιώνει και για την, ε, επανεγκα... μετεγκατάσταση. Υπάρχουν πολλές συζητήσεις γι' αυτό. Πότε νομίζετε όμως ότι θα πρέπει να αναλυφθεί δράση κατά των κατομέλων που δεν σέβονται την νομοθεσία την οποία τα ίδια ανέκριναν. Για το πρώτο μέρος της ερώτησής σας έχει να κάνει με το δεύτερο σημείο για την επανεκατάσταση, την μετεγκατάσταση. για την ώρα η μετεγκατάσταση ε, λειτουργεί. Οπότε δεν θα αντιμετωπίσουμε τέτοια δυσκολία. Αλλά θα πρέπει να είμαστε επανέτοιμοι. Ο αριθμός που αναφέρατε προηγουμένως είναι ένα πρώτο στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη για να δικαιολογηθούν ε, τα κινητρά μας. Ως προς τη δεύτερη παράμετρο του ερωτήματός σας, το γνωρίζουμε. Και έχουμε τα πρώτα θετικά δείγματα το τελευταίο καιρό, το τελευταίο διάστημα, με την κατάσταση και εκεί να λειτουργεί. Έχει αρχίσει να φέρνει αποτελέσματα το σύστημα και έχουμε περίπου 6.000 άτομα τα οποία μετεγκαταστάθησαν πρόσφατα. Άρα αρχίζει να λειτουργεί. Βεβαίω δεν τα έχουμε καταφέρει ακόμη και όντω δεν θα κρύψω και εγώ την απογοήτευσή μου για το γεγονό ότι το τελευταίο διάστημα πολλά κρατημέλη δεν ανταποκρίθηκαν θετικά στι ε, δεσμεύσει του. Όμω η κατάσταση έχει βελτιωθεί πολύ. Πιστεύω προσωπικώ ότι είναι θέμα χρόνου προκειμένου το πρόγραμμα μεταγκατάσταση να λειτουργήσει σε όλα τα επίπεδα. Και βεβαίω αυτό με φέρνει πάλι πίσω στο πρώτο τμήμα τη ερώτησή σα τον αριθμό, τον αριθμό αυτών των ανθρώπων που δεν θα μείνουν στην Ελλάδα, ΕΣΑΗ. Ευχαριστούμε. Άλλος κανείς, παρακαλώ. Uh, Ήθελα να μάθω πόσο καιρό μπορείτε ακόμα να παρατείνετε αυτό το μέτρο πέραν των τριών μηνών. Μπορείτε τεχνικά να παρατείνετε και για άλλους δύο μήνες και πόσες φορές και για πόσο. θέλετε να δείτε ε, ποιο, ε, ποιος θα είναι η χρονική περίοδος της παράτασης. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι εργαζόμαστε πάνω στο θέμα αυτό από τον περασμένο Μάρτιο και το γεγονός ότι είμαστε σε θέση σήμερα να δώσουμε μια θετική απάντηση στο αίτημα ε, που υπέβαλαν αυτά τα κράτη-μέλη δεν σημαίνει ότι η παράταση θα διαρκέσει επάπειρον. Θα επαναλαμβάνεται. Ο χρόνος ε, που έχουμε ενώπιόν μας είναι πάρα πολύ περιορισμένος. Τέσσερις, ε, τρεις μήνες είπαμε. Πιστεύω ότι στο τέλος αυτής της τρίμηνης περίοδου, εάν υπάρχουν δικαιολογημένοι λόγοι, ε, θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι, αλλά πιστεύουμε ότι αυτοί οι τρεις μήνες θα είναι το τέλος της περίοδου και ότι θα επανέλθουμε στη φυσιολογική κατάσταση ε, και ότι θα μπορεί να λειτουργήσει πλήρως το σύστημα Schengen. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, υποστηρίζετε την απόφαση των γαλλικών αρχών να καταστρέψουν, να εξαλείψουν τη ζούγκλα του Καλέ από τη στιγμή που η εκένωση ε, της ζούγκλας, της λεγόμενης ζούγκλας, λαμβάνει χώρα με συνθήκες που δείχνουν σεβασμό απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Υποστηρίζουμε αυτήν την πρωτοβουλία και από ό,τι ξέρουμε η επιχείρηση επιτόπου γίνεται με πλήρη σεβασμό των δύο αρχών που ανέφερα προηγουμένως. Αναμενόταν να συμβεί αυτή η εκένωση και νομίζω ότι οι γαλλικές αρχές τώρα υλοποιούν αυτό που έχουν αποφασίσει με πλήρη ευθυγράμμιση και τήρηση των ε, αντιλήψεων των αρχών που ανέφερα. Θα ήθελα να επανέλθω στην προηγούμενη ερώτηση, διότι από ό,τι καταλαβαίνω ε, δεν ήταν σχετικά με το χρόνο, με την χρονική περίοδο. Ρωτήσατε επίσης τι θα συμβεί μετά τους τρεις μήνες. Αν κατάλαβα σωστά αυτό το οποίο είπατε. Μέχρι πότε, μέχρι πότε είπατε. Αυτό με ρωτήσατε προηγουμένως. Ναι, ναι. Διότι θα ήθελα να επανέλθω. Μπορείτε να επαναλάβετε την ερώτησή σας Νομίζω ότι ήταν για την τελική χρονική περίοδο μετά από αυτούς τους τρεις μήνες. Πόσες παρατάσεις μήνες Θα ήθελα να διευκρινίσω το θέμα. Το Συμβούλιο, διότι αυτή η πρόταση υποβάλλεται στο Συμβούλιο, όπως ξέρει, μπορεί να παρατείνει την αρχική περίοδο όχι περισσότερο από τρεις φορές μέχρι μία περίοδο έξι μηνών και το μέγιστο θα είναι δύο χρόνια εάν υπάρχουν εξαιρετικές περιστάσεις που να συνεχίζονται. Αν αυτή είναι η περίπτωση, θα αποτιμήσουμε την κατάσταση και θα εξετάσουμε εάν οι λόγοι αυτοί είναι πλήρως δικαιολογημένοι. Τα δύο χρόνια που ανέφερα προηγουμένως αποτελούν μια δυνατότητα βάσει του άρθρου 29. Μια δυνατότητα. Και θα ήθελα να το διευκρινίσω αυτό δεν είναι μια υποχρέωση. Το Συμβούλιο μπορεί να παρατείνει για λιγότερο από την συνολική περίοδο των δύο ετών. Βεβαίως, ο στόχος, όπως είπα στην αρχή, είναι να επανέλθουμε σε μια φυσιολογική λειτουργία του Σέγγεν και να μην εξαντλήσουμε ε, τα έξι χρόνια. Δα τα δύο χρόνια, με συγχωρείτε. Από το Bloomberg, για αυτό το σημείο για να είναι σαφές περιμένετε ότι σε τρεις μήνες μπορεί να επανέλθει πλήρως το Σέγγεν, αλλά δεν το ξέρουμε ακόμη. Θα ήταν λογικό να υποστηρίξουμε ότι προτείνοντας μόνο μία τρίμηνη περίοδο, αντί για τη συνήθη περίοδο έξι μηνών, δεν ε, απεκδίεστε τις δυνατότητε να αξιοποιήσετε και τα δύο χρόνια. Δεν χάνετε τους τρεις μήνες από τα έξι χρόνια. Μπορείτε να επανέλθετε ο κύριος Αβραμόπουλος. Ε, εξήγησα ποιες είναι οι δυνατότητες εάν υποβληθεί νέο αίτημα στο μέλλον. Αλλά ήμουν και πολύ σαφής για το στόχο μας. Ο στόχος μας είναι να επανέλθουμε σε ένα πλήρως λειτουργικό Σέγγεν. Ρίκ Rinkle. Αυτή η παράταση μοιάζει να σχετίζεται άμεσα με την κατάσταση στην Ελλάδα. Δώσατε στις ελληνικές αρχές περίοδο τριών μηνών για να βελτιώσει την κατάσταση στα hot spot και να, επιστρέψουν, να αρχίσουν να επιστρέφουν στην Τουρκία. Οι ελληνικές αρχές έχουν πάρει πολλά έψημα για τις επιδόσεις τους τους τελευταίους μήνες. Είναι αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει υπερβολικός φόρτος στην Ελλάδα που έχει μείνει από προηγουμένως όμως μας έχουν δοθεί διαβεβαιώσεις από τις ελληνικές αρχές ότι πολύ γρήγορα οι αιτήσει ασύλου θα τύχουν επεξεργασίες πολύ γρηγορότερα ώστε οι επιστροφές προς την Τουρκία θα λάβουν χώρο στο δυνατόν συντομότερα. Διότι αυτό είναι το, αυτή είναι η μεγάλη αδυναμία των επιτόπου διαδικασιών αυτή τη στιγμή. Ω προ τα λοιπά, όλα πηγαίνουν, ε, βαίνουν καλώ. Ε, είναι αλήθεια, όπω είπα και στην αρχή, ότι ο αριθμό αυτό των ανθρώπων δεν θα παραμείνουν μέσα στην Ελλάδα. Οι ελληνικέ αρχέ κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Βεβαίω με την πλήρη στήριξη των υπηρεσιών μα και γενικότερα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι η κατάσταση όσο έχει σήμερα και ελπίζω ότι η κατάσταση όσο έχει σήμερα δεν θα συνεχιστεί του επόμενου μήνε, αλλά να επανέλθω στο αρχικό ερώτημα. Όχι. Δεν θα στείλουμε τελεσίγραφο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, διότι κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Του βοηθούμε, του στηρίζουμε και πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα η κατάσταση θα ε, εξομαλυνθεί πλήρω. Ακόμη και στο επίπεδο των διαδικασιών που θα πρέπει να ακολουθούν οι τον άσυλο. Ευχαριστούμε, Επίτροπε. Σας ευχαριστώ όλους. Καλό σας βράδυ.